Σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθίστε. Άρχεται η συνεδρίαση. Σας παρακαλώ να καθίσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνεται τη συνεδρίαση. Έχω διάφορα τεχνικά πρώτα να σας ανακοινώσω. Να σας πω ποιες είναι οι πολιτικές ομάδες που σχηματίστηκαν στο Κοινοβούλιο. Είναι το κόμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ε, Χριστιανοδημοκράτες, η κοινοβουλευτική ομάδα που αριθμεί 221 μέλη. Στη συνέχεια, Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, S&D, η σύντμηση έχει 191 μέλη. Η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ECR, 70 μέλη. Η ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, σύντμηση 67 μέλη η Συνομοσπονδιακή Ομάδα Ενωτικής Αριστεράς και Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, GUE-NGL, 52 μέλη. Η Ομάδα των Πρασίνων και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας, ΒΕΡ, Ale 50 μέλη. Και η Ομάδα της Ευρώπης Ελευθερίας των ελευθεριών συγγνώμη, και της άμεσης δημοκρατίας η FTD με 48 μέλη. Μία εγγεγραμμένη ε, παραμένουν 58 ευρωβουλευτές. Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 του κανονισμού διαβιβάζονται στον Πρόεδρο ε, οι δηλώσεις για την συγκρότηση αυτών των ομάδων και ανακοινώνονται ούτως στο σώμα. Οι αρμόδιες Ιταλικές αρχές ενημέρωσαν το Κοινοβούλιο από 18 Ιουνίου για την εκλογή του κυρίου